Good afternoon to all of you and uh, especially to our colleagues. Καλησπέρα και ιδιαίτερα ε, καλησπέριζουμε τους συναδέλφους από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Πολύ λυπάμαι για την ε, καθυστέρηση. Δεν είστε. Δεν είναι γερμανικός τρόπος ε, διεξαγωγής μιας συνεδρίασης. Ξέρω ότι οι Γερμανοί συνάδελφοι θα ήταν εδώ στην ώρα του και θα ξεκινούσαμε στην ώρα μα, αλλά αυτή είναι η Ευρώπη, αυτέ είναι οι Βρυξέλλε. Καλώ ορίσατε και θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία πρωτού μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Αλλά τώρα, 15.06 πλέον, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μα. Το πρώτο θέμα Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει στην ημερήσια διάταξη, μπορεί να εγκριθεί. Θεωρώ ότι είναι εγκεκριμένη λοιπόν η ατζέντα. Then I have a few announcements. Έχω μερικέ αναγγελίε. Σα ενημερώνω ότι η δημόσια ακρόαση για την πρωτοβουλία για τους, των Ευρωπαίων πολιτών θα γίνει Δευτέρα 11 Μαΐου από τις 3 έως 6.30 το απόγευμα. Αυτή η ακρόαση οργανώνεται από την Επιτροπή Γεωργίας μαζί με εμά, με την Επιτροπή ΕΜΒΗ και με την Επιτροπή ΙΤΡΕ. Και θέλω να σας ενθαρρύνω όλους να παραστείτε στην ακρόαση αυτή και να ενημερώσετε και τη γραμματεία εκ των προτέρων, εάν θα συμμετάσχετε, ούτω ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή οργάνωση σε ό,τι αφορά το χρόνο και τα διαδικαστικά. Λοιπόν, αφού διεκπαιρεώσαμε αυτό, πάμε στο σημείο 3. Διάφορα, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Και τώρα με μεγάλη χαρά θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους και φίλους από την Επιτροπή Αναφορών της Γερμανικής Bundestag. Εδώ στο βήμα έχω την κυρία Στάνκε που είναι η πρόεδρος της δικής σας Επιτροπής της Bundestag. Είχαμε και θα έχουμε επικοδομητική συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων και εμπειρίες επιμερισμό βέλτιστων πρακτικών κτλ. Και μετά από αυτή την ανταλλαγή απόψεων, η Επιτροπή μας θα εξετάσει μια σειρά αναφορών από τη Γερμανία ή αναφορές που αφορούν τη Γερμανία. Τη μία σας την ε, προωθήσαμε και ελπίζω να σας φαίνεται ενδιαφέρουσα. Και θα δείτε και πώς ε, ασχολείται και πώς διεκπαιρεώνει η Επιτροπή μας έτσι, αυτές τις αναφορές από πρώτο χέρι. Πριν να συζητήσουμε τα κοινά μας θέματα, που είναι φυσικά οι αναφορές, θα ήθελα επευκαιρία να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών, όλους σας από την Γερμανική Bundestag και τα μέλη του προσωπικού και τη Γραμματεία για την ε, υποστήριξή τους πέρυσι και φέτος. Πέρυσι δεν ήμουν εγώ πρόεδρος, αλλά... Αλλά είμαι σίγουρη ήταν επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Πέρυσι η δίκηση έκανε μία μελέτη για τον τρόπο που διεξάγονται οι αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για να μάθουμε από την εμπειρία που έχουν άλλα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, οι συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα μέλη της γραμματείας τα προσκαλέσαμε. Η... Το προσωπικό μας πήγε στη Γερμανία και είδε πώς δουλεύετε και έτσι εμπνεύστηκε με διάφορες ιδέες για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής μας. Στο μέλλον θα μπορούσαμε να ανταλλάσσουμε απόψεις για να χρησιμοποιούμε με καλύτερο τρόπο τι αναφορές στην νομοθετική διαδικασία. Δηλαδή, με τρόπο τους ώστε να συνεργαζόμαστε ακόμα περισσότερο με τις νομοθετικές επιτροπές και αρμόδιες γενικά επιτροπές στου διάφορου τομεί αρμοδιότητας του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει επίσης να ανταλλάσσουμε απόψεις για θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέματα που αφορούν τοπικές ή περιφερειακές αρμοδιότητες επίσης. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να μάθουμε από εσά από τη Γερμανική Επιτροπή Αναφορών. Σας ευχαριστώ εγώ προσωπικά, ε, τα μέλη της Γραμματείας και οι συνάδελφοι που ήρθαν εδώ για να συζητήσουμε μαζί σας και θα σας υποστηρίξουμε και εμείς με τον ίδιο τρόπο, εάν παρελπίδα το χρειαστείτε. Μην, έχετε, μην διστάσετε να μας υποβάλλετε ερωτήματα να μιλήσω λιγάκι για τα δικαίωμα των αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με βάση το άρθρο 227 της Συνθήκης και το άρθρο 44 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, κάθε Ευρωπαίος πολίτης και κάθε κάτοικος μπορεί να υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα που αφορούν του τομεί τη δραστηριότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή Αναφορών ε, εργάζεται και σας διαβεβαιώ ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διερευνήσουμε θέματα που θέτουν οι αναφέροντες. Πέρυσι, το 2014, η Επιτροπή μας έλαβε 2.719 αναφορές. Είναι πολλές. Τις περισσότερες αναφορές τις αφορούν θέματα περιβάλλοντος, εν συνεχεία θέματα θεμελιώδη δικαιώματα και θέματα ενίας αγοράς, δικαιοσύνη και θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και αυτά τα θέματα αφορούν τις αναφορές μερικές φορές, καθώς και θέματα που αφορούν τα οικονομικά θέματα, χρηματοπιστωτικά και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Είμαστε υπεύθυνη επιτροπή επίσης για τις σχέσεις με τον Ευρωπαίο Δημασουλαβητή και οργανώνουμε την εκλογή του διαμεσολαβητή. Παίζουμε σημαντικό ρόλο επίσης στην πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτειών. Συνδιοργανώνουμε δημόσιες ακροάσεις για αυτό το θέμα ε, που αφορά τις ε, πετυχημένες πρωτοβουλίες. Είναι αυτές οι οποίες έχουν τουλάχιστον εκατομμύριο υπογραφές σε 7 διαφορετικά κράτη-μέλη. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά για αυτά που κάνουμε, αλλά είμαι σίγουρη ότι τα έχετε μελετήσει πριν έρθετε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν <clears throat> θα ήθελα να τονίσω κάτι που μας κάνει ιδιαίτερα περήφανος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε σημειώσει πρόοδο από τη στιγμή που εισάγαμε το web streaming στις συνεδριάσεις μας. Αυτό επιτρέπει στους πολίτες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα 28 κράτη-μέλη, να παρακολουθούν τις συζητήσεις στην Επιτροπή μας για θέματα που αφορούν τις αναφορές τους και αν δεν μπορούν να παραστούν βέβαια τις παρακολουθούν μέσω του ίντερνετ ο, ή ε, παρακολουθούν σε περίπτωση που τους ενδιαφέρει ο τομέας. Επίσης υπάρχει και μια νέα δικτυακή πύλη που θα είναι πολύ χρήσιμη στο μέλλον. Αυτή η πύλη δίνει πληροφορίες και τον τρόπο για να υποβάλει κανείς αναφορά. Εξηγεί πώς υποβάλλεται μια τέτοια αναφορά. Μπορεί να δει κανεί ε, σε τι φάση είναι η αναφορά του και τι θέματα καλύπτουμε στου διάφορου τομείς δραστηριοτήτων μα. Η επιτροπή σας ήταν μία από τις ε, βασικές επιτροπές στην Bundestag στις επιγραμμικές αναφορές. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να μάθουμε από τις εμπειρίες σας σε αυτόν τον τρόπο ανταλλαγής απόψεων τον επιγραμμικό δηλαδή, μέσω ίντερνετ. Επίσης θέλουμε να δούμε πώς ε, διεκπεραιώνουμε εμείς και εσείς. Ε, αν τις αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο ή αν υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των πολιτών. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για το πώς θα διευρύνουμε ή θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Και με ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος προς αυτήν την κατεύθυνση να μου πείτε εάν η μορφή ενός δικτύου με την Επιτροπή Αναφορών ή Επιτροπή Αναφορών στην Ευρώπη και φυσικά τη δική μας Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν ιδέα ενός δικτύου αξίζει τον κόπο να την ψάξουμε. Συνολικά, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι τα κοινοβούλια εκλέγονται για να εξυπηρετούν και να υπηρετούν τους πολίτες και να προωθούν τα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης. Αυτό ε, εξυπηρετείται μέσω των διαδικασιών και των λειτουργιών των Επιτροπών Αναφορών ή της πρωτοβουλία για τους πολίτες, ε, μέσω των θεμάτων που οι ίδιοι οι πολίτες μας υποβάλλουν και που αξίζει να εγκύπτουμε σε αυτά. Είναι χαρμόσυνη μέρα λοιπόν σήμερα και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον στην επικεφαλή τη Γερμανική αντιπροσωπείας, την κυρία Στάνκε. Έχετε το λόγο. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε Βίξτρομ, αξιότιμοι συνάδελφοι, καταρχά θα ήθελα να σα ευχαριστήσω να ευχαριστήσω τον ε, Δόκτωρα Γιάννη και τον ε, κύριο Βίλαν που μας ενημέρωσαν για τον τρόπο λειτουργία της Επιτροπής, της Επιτροπής Αναφορών. Να ευχαριστήσω και τους υπαλλήλους της Επιτροπής σας. Ε, χαιρόμαστε που βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε μαζί θέματα και την επεξεργασία των αναφορών. Συνεχίζουμε τον διάλογο από την τελευταία θητεία και από εδώ τι είχε φανεί πόσο απαραίτητο είναι να γνωρίζουμε τις εργασίες και τον τρόπο λειτουργίας των άλλων επιτροπών. Στη Γερμανία αυτό τι συμβαίνει, ότι η επεξεργασία των αναφορών γίνεται σε επίπεδο ομοσπονδιακό, αλλά και ομόσπονδο επίπεδο κρατηδίων. Και έτσι έχουμε λοιπόν σαφά, σαφώς αρμοδιότητε. αρμόδιοτητες. Είτε λοιπόν είναι αρμόδια η Ομοσπονδία, το Ομοσπονδιακό κράτο, είτε τα κρατήδια. Υπάρχει λοιπόν ε, σαφή διαχωρισμό στη Γερμανία. Και κάθε επίπεδο είναι υπεύθυνο και αρμόδιο μέχρι τη τελική ε, επεξεργασία. Κανείς δεν μπορεί να υποβάλει ένσταση αν δεν έχει αρμοδιότητα. Εμάς μας απασχολεί τουλάχιστον πιο πολύ το επίπεδο το ευρωπαϊκό σε σχέση με το εθνικό κυρίως και το πώς μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω η επικοινωνία και η διαπαφή και κατά πόσον μπορούμε να έχουμε ένα πρότυπο ένα πρότυπο όπως αναφέρετε και εσείς κυρία Πρόεδρε. Ο διαρκής διάλογος όμως είναι απαραίτητος γιατί οι εμπλεκόμενοι φορείς, τα άτομα στην Επιτροπή μας, ο κύριος Στόερχαν, ο συνάδελφος Μπάουμαν, νομίζω ότι είναι οι μοναδικοί που ήμασταν ε, εδώ στην τελευταία συνάντησή μας. Η Επιτροπή Αναφορών θεωρώ ότι είναι ο σεισμογράφος του Κοινοβουλίου και εδώ βλέπουμε πώς επιτρούν οι νόμοι στους πολίτες. Σε καμία άλλη επιτροπή κοινοβουλευτική δεν έχουμε τόσο άμεση εκπροσώπηση των ενστάσεων, των παραπώνων των πολιτών. Είτε πρόκειται για θέματα υγείας, συντάξεων, είτε πρόκειται για ένα δυστύχημα όπως αυτό της Φοκουσίμα, οι πολίτες απευθύνονται στην Επιτροπή Αναφορών πάντα σε εμά, του βουλευτές. Και προσπαθούμε εμείς να βοηθήσουμε. Και συχνά ασχολούμαστε πιο πριν με, από τις αρμόδιες επιτροπές με τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο. Αλλά είναι και, αν θέλετε, μια κάρτα επισκέψεων η Επιτροπή Αναφορών σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο. Δείχνουμε δηλαδή στου πολίτε πώ αντιμετωπίζουμε τι ανησυχίε του τα προβλήματά του. Επιτρέψτε μου να θέσω τρει κατευθυντήριε γραμμέ για τι εργασίε μα. Καταρχά, μη μονομένη βοήθεια, αν οι πολίτε έχουν αδικηθεί. Δεύτερον, η λειτουργία απόπειρα συμφιλίωση των πολιτών με την κατοική απόφαση, αν δεν είναι δυνατόν να τερθωθεί αυτή. Και τρίτον, νομοθεσία που θεωρεί ο πολίτης ότι τον έχει πλήξει ιδιαίτερα κρίσιμο κρίνω το θέμα της δεύτερης λειτουργίας αυτής, της ικανοποίησης των πολιτών. Δεδομένης της ε, υφιστάμενης νομοθεσίας. Δεν αρκεί απλά να πούμε στον ε, αναφέροντα τι ισχύει. Εμείς ε, πρέπει να καλέσουμε τον πολίτη να συμφιλειωθεί με την πραγματικότητα. Και μπορεί να μην μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά συνήθω όταν οι πολίτες μας ευχαριστούν για τις σωστές και πλήρες εξηγήσεις, ξέρουμε ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά. Και αυτό προωθεί τους πολιτικούς θεσμούς. Δεν είναι απλό το έργο, αλλά πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντά μας. Εξαιρετικά επίκαιρο και πρέπει να είμαστε ευγνώμονε όταν απευθύνονται σε εμά οι αναφέροντα. Δείχνει ότι οι πολίτε συμμετέχουν στο πολιτικό γίγνεσθε, ότι έχουν εμπιστοσύνη σε εμά του πολιτικού. Και πρέπει λοιπόν να σταθούμε και να αποδεχτούμε αντάξει τη εμπιστοσύνη αυτή. Η Επιτροπή μας λαμβάνει 16.000 ε, αναφορές κάθε χρόνο. 20% αφορούν τα εργασιακά και τα ελληνικά θέματα και 10% τα Υπουργεία Ιστορικών, Δικαιοσύνης, Προστασίας Καταναλωτών και Οικονομικών. 15% δεν εμπίπτει στο μου διαθετά μα. Και αν είναι κάποια άλλη επιτροπή αρμόδια ή κάποιο άλλο σώμα αρμόδιο, το προωθούμε την αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στο ομόσπονδο επίπεδο, ομοσπονδιακό επίπεδο. Δύο είναι οι βουλευτές που ελέγχουν ε, από πλευρά ε, τη κυβέρνηση και από πλευρά τη αντιπολίτευση στην ε, κάθε αναφορά και τελικά η Ολομέλεια κυβερνηση και απο πλευρα τη αντιπολιτευση την καθε αναφορα και τελικα η ολομελεια αποφασιζει για το κατά πόσο είναι παραδοκτή η αναφορά. Και επειδή υπάρχει αυτή ο διαχωρισμός ε, αρμοδιοτήτων, μπορούμε να αποφθενόμαστε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, το οποίο ενδεχομένω να φαίνεται ότι είναι ατελές, αλλά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση με την ε, μεταφορά μιας αναφοράς μπορεί να πετύχει καλύτερη επεξεργασία της. Και συχνά είναι πολλοί αυτοί οι αναφέροντας, οι οποίες ανεξάρτητα το ένα από τον άλλον ε, υποδεικνύουν την ίδια, το ίδιο πρόβλημα. Εδώ πέρα λοιπόν η Επιτροπή Αναφορών προτείνει ένα διαφορετικό μηχανισμό. Με μεγάλη επιτυχία από το 2005 έχουμε και τον κόμβο αναφορών που είναι ηλεκτρονικός. Έχει στη μεγαλύτερη επιτυχία περίπου 40% λοιπόν όλων των αναφορών καταφτάνουν με τον τρόπο αυτό. Και έχουμε πάνω από 1,8 εκατομμύρια χρήστες. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο έχει επιτυχία ο κόμπος αυτός, η πύλη αυτή, αλλά ότι μέσω αυτού ενημερώνουμε και αγγίζουμε πιο πολλούς πολίτες. Μία ερώτηση και μία παρατηρήση, επιτρέψτε μου. Τι θα κάνει η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου με τις αναφορές που του διοχετεύουμε, ίσως θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε ένα σύστημα feedback. Αυτό θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για τις εργασίες μας. Αν ξέρουμε δηλαδή το τι κάνετε τελικά με τις ε, αναφορές που σας δώσαμε και η παρατήρηση. Ως τώρα ήταν πολύ επίσημη η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Χρονοβόρα, διαδικασία και κοστοβόρα. Θα μπορούσε να υπάρξει μια απλούστευση, να υπάρχει άμεση επικοινωνία σε επίπεδο εργασία. Με τα κρατήδια στη Γερμανία έχουμε μια πιο απλή διαδικασία η οποία λειτουργεί εξαιρετικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ θα σταματήσω και άλλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα επεξηγήσουμε στις περαιτέρω συζητήσει με τους συναδέλφους από την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στα μέλη για τη συζήτηση. Να περάσω πρώτα στους συντονιστές ε, των επιμέρους ομάδων. Πίτερ, θες να πάρεις πρώτα το λόγο. Να ξεκινήσω έχω και συγκριτικό πλεονέκτημα γιατί είχαμε κάνει ήδη μια πρώτη συζήτηση πριν από λίγο με του συναδέλφους από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Σα καλώς ορίζω εκ πάτους καρδιά, Πολύ καλή εισαγωγή και κατέδειξε πώς έχουν τα πράγματα κοντά στον κόσμο είπατε. Είπατε ότι είμαστε σεισμογράφος ε, των πολιτών και εμείς έτσι θεωρούμε ότι λειτουργούμε και πιστεύω ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι η η Επιτροπή η οποία είναι ενημερωμένη για το τι συμβαίνει και ποια είναι τα συναισθήματα που επικρατούν στον κόσμο. Δύο παρατηρήσεις επιτρέψτε μου. Έχουμε ασφαλώς τον ίδιο στόχο. Το δυνατόν γρήγορότερα να επεξεργαζόμαστε τις αναφορές. Και είναι και καλή η κατανομή των αρμοδιοτήτων. Έχουμε λοιπόν ε, νομοθετικές προτάσεις, είπατε, και εμείς το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε το θέμα της ικανοποίησης των πολιτών ε, είναι κάτι που μας απασχολεί και εμάς σε ό,τι αφορά τους αναφέροντας. Πάντα με εντυπωσιάζει το γεγονός όταν λέμε ότι γίνεται γοργή ανταλλαγή και διοχέτευση των αφορών για να γίνεται και η γουργή διεκπαιρίωσή του. Γιατί όσο καθυστερούμε, τόσο κάτι χάνεται. Το επόμενο θέμα που ήθελα να θέσω το είπε και η πρόεδρος Βίξτρεμ. Ξέρουμε ότι στις καθημερινές μας ε, λειτουργίες υπάρχουν ελαττώματα και έλλειμματα. Θέλουμε λοιπόν να αναπτύξουμε ένα δίκτυο αναφορών. Πώς το βλέπετε εσείς, ε? πιστεύετε ότι υπάρχει σκοπός, υπάρχει λόγος να συνεχίσει αυτή η ανάπτυξη δικτύου. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο τον λόγο, το οποίο με ικανοποιεί γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Κύριε Μαχτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πάω κατευθείαν στο ψητό. Αν μου επιτρέπετε, όπως είπα και η κυρία Πρόεδρο πολύ σωστά, είμαστε εδώ για να εκπροσωπήσουμε και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα όλων των πολιτών. Εφόσον απευθύνομαι με μεγάλη μου χαρά σε ένα μέλος της θα έχω τρία ερωτήματα για το Jugendamt. Εδώ είμαστε στην Επιτροπή Αναφορών, λαμβάνουμε πάρα πολλές αναφορές και πολλές από αυτές, από πολλούς Ευρωπαίους πολίτες, λένε ότι έχουν πέσει θύμα της Jugendamt. Και εγώ προσωπικά έχω αναλάβει 10 τέτοιες αναφορές. Ελπίζουμε να τις ε, εξετάσουμε τίματα την άλλη. Τρία συγκεκριμένα ερωτήματα να σας θέσω. Έλαβα πολλές σελίδες ε, ερωτήσεων, αλλά δεν έχει νόημα να τα θέσουμε όλα αυτά. Τα τρία πιο εύστοχα ερωτήματα. Πρώτον, γιατί η Γερμανία χρησιμοποιεί μια τέτοια διοικητική διαδικασία, Battenstaft, ε, που κάτι που υπερισχύει από το οικογενειακό δικαστήριο, ε, κάτι το οποίο προδικάζει πολλές φορές, ε, προκαταλαμβάνει και τις μελλοντικέ διαδικασίες στο αστικό δικαστήριο. Γιατί είναι διοικητική δομή το Jugendamt πώς μπορεί να επιτυχεί. Και τρίτον, πώς ένας ο μη Γερμανός μπορεί να ε, αποδείξει ότι για το παιδί του ε, που έχει πολύ καιρό να το δει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να το απαγάγει. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που βρίσκονται σε δραματική κατάσταση, εδώ και πολλά χρόνια δεν έχουν το δικαίωμα να επισκεφθούν και να δουν τα παιδιά τους. Δεν έχουν δικαίωμα επίσκεψη λοιπόν. Περιμένω τις απαντήσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ η Ελεονόρα Εύη. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να υποφεληθώ από την ευκαιρία που έχουμε. Για να υποβάλω καταρχάς ένα ερώτημα. Ο αριθμός των αναφορών που λαμβάνεται σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα. Δεν κατάλαβα. Ίσως το έχασα το σημείο αυτό που είπατε. Τι είδους αναφορές λάβατε, πόσες αναφορές λάβατε. Νομίζω ότι ε, είναι πολύ δυσανάλογες οι αναφορές που είπατε ότι λαμβάνετε εσείς για το περιβάλλον σε σχέση με αυτές που λαμβάνουμε εμείς. Έπειτα, όπως και στον με αυτά, θέλω να υποβάλω ένα ερώτημα που συνδέεται περισσότερο με την ποσότητα αναφορών. Λαμβάνετε αναφορές ε, για αυτό το δικαστήριο ανηλίκων, το Jugendamt. Γιατί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, λαμβάνουμε πάρα πολλές αναφορές. Πολύ συχνά δεν καταφέρνουμε ούτε καν να δώσουμε πλήρεις απαντήσεις. Υπάρχουν καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες. Η Bundestag λαμβάνει αναφορές για αυτό το θέμα το δικαστήριο υλίκων. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ήθελα αρχικά ε, να στηρίξω όλες τις αναφορές που συνδέονται με το Jugendamt, αλλά όχι μόνο ε, για τις γερμανικές αρχές, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο τη Γερμανία. Είναι ένα γενικό ζήτημα, το οποίο βλέπω ως εξής απομακρύνουμε τους γονείς από τα παιδιά τους. Είναι μια παράνοια που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Κάποιες φορές για σήμαντους ε, λόγους, ανυπόστατους μάλιστα. Είναι βάναυση αυτή η πρακτική και δημιουργεί σημαντικά προβλήματα και ψυχολογικά και για τα παιδιά. Εγώ αντιτάσσομαι σε αυτή την ε, πρακτική. Από την άλλη, βλέπουμε ότι πρόκειται για ε, πρακτικές που, που χρηματοδοτούνται και από το κράτος και δεν λαμβάνουν υπόψη καν τα συμφέροντα των πολιτών και την ευημερία τους. Το έχω εξετάσει σε πολλές περιπτώσεις. Ε, ομολογώ ότι ορισμένες φορές έχω την εντύπωση ότι είναι σαν μια υπόθεση, μια ένα δίκτυο που θυμίζει μαφία. Απομακρύνονται κάποια παιδιά από ορισμένε οικογένειε που δεν έχουν ε, που δεν υπάρχει παθολογική κατάσταση. Και έτσι, ακόμα και όταν δεν υπάρχει πρόβλημα, όταν έχουμε μια ε, οικογένεια που είναι υγιής και λειτουργεί μια χαρά και πάλι βλέπουμε ότι απομακρύνονται τα παιδιά από εκεί. Είναι λοιπόν μια τρέλα που υπάρχει στην Ευρώπη και σίγουρα υπερβαίνει τα εύλογα όρια. Εγώ έχω ε, δει με τα μάτια μου πολλές οικογενειακές τραγωδίες που οφείλονται σε αυτό. Γι' αυτό στηρίζω όλες τις αναφορές που συνδέονται με αυτό το ζήτημα. Πρέπει να κάνουμε κάτι στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε κάποιος από την Πούντες να λάβει το λόγο. Yes. Oh, sorry, I didn't see you. Α, συγγνώμη. Η κυρία Στανόκα πρώτα. And please, if anybody from Bundestag... Και μετά αν θέλει κάποιο να πάρει το λόγο την Bundestag. Yeah, one more question. Ακόμα μία ερώτηση. Μια και οι συνάδελφοι θέσαν το θέμα της Jugendamt. Υπάρχει θέμα όπου επλέκονται περισσότερα από ένα κράτη. Συνήθως, ειδικά όταν φτάνουν αυτές οι αναφορές ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από μεικτά ζευγάρια συνήθω, από μεικτού γάμου. Εξετάσαμε μια υπόθεση είχαμε μία αναφορά από τη Γερμανία που αφορούσε περιβαλλοντικά θέματα, αφορούσε ε, ορυχεία στο που επηρεάζονται από τους καταράχτες. Η εταιρεία ήταν σουηδική. Έγινε μια οικολογική καταστροφή εκεί. Έχετε κάνει ακροάσεις. Εγώ προσωπικά ασχολήθηκα με αυτό το θέμα πριν από δύο εβδομάδες. Λάβατε τίποτα εσείς κάποια αναφορά για το θέμα αυτό ε, και την έχετε διεκπαιρεώσει. Ευχαριστούμε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην ε, κυρία Μπορμπέκη Κάισερ. Σας ευχαριστώ για το πώς η Γερμανία αντιμετώπισε το θέμα του, δικαίωμα, του δικαιώματος, ε, της αφαίρεσης του δικαιώματος ε, εποπτείας και κυδαιμονίας ανελίκων. Είναι πολύ ψηλά το εμπόδιο προτού αφαιρεθεί το δικαίωμα αυτό της κυδαιμονίας από το γονιό. Και στη Γερμανία γίνεται η ευθεσία μόνο αν οι γονείς συμφωνήσουν. Ή αν υπάρχει συμφωνία το γονιού, αν του έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα κυδαιμονίας και το παιδί βρίσκεται σε ίδρυμα ή σε αυτή την οικογένεια. Η οθεσία υπάρχει μόνο με την έγκριση των γονέων. Και έτσι λοιπόν στο Γερμανικό Κοινοβούλιο είναι λίγε οι περιπτώσει που φτάνουν σε εμά, γιατί είναι η συντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων λύνεται στα δικαστήρια ή στο Jugendamt. Ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη χαρά θα δώσω τώρα το λόγο στους τη Γερμανίδα ομολογό μου για να απαντήσει τις ερωτήσεις που υποβάλατε. Εν συνεχεία θα μπούμε στις αναφορές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα μέλη της Bundestag θα δουν πώς εμείς ε, ασχολούμαστε με τις αναφορές αυτές. Το θέμα για το Jugendamt το απάντησε στην συνάδελφος. Υπάρχουν λοιπόν σαφώς ορισμένες αρμοδιότητες Υπάρχουν θέματα που είναι αρμοδιότητα των ομόσπονδων κρατηδίων, υπάρχουν θέματα που είναι αρμοδιότητα του ομοσπονδιακού κράτου. σε ό,τι αφορά τις θέματα περιβάλλοντο. Δεν μπορώ να σα δώσω αριθμητικά στοιχεία, αλλά ασφαλώ τα επεξεργάζεται όπως αρμόζει η Επιτροπή μας. Υπάρχει και μια ετήσια έκταση και στα αγγλικά που μπορούμε να σας διαβιβάσουμε σε ό,τι αφορά το δίκτυο των Επιτροπών Αναφορών. Είμαι πάρα πολύ ανοιχτή προς αυτό. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διαμεσολαβήσεων για τις αναφορές. Συμμετέχει και το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ καλή λοιπόν η συνεργασία στο επίπεδο αυτό. Αλλά βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα της δικτύωσης η συνεργασία αυτή είναι πολύτιμη, την καλωσορίζω. Και κάποιο θα πρέπει να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία, μάλλον από πλευρά τη Ευρώπη, υποθέτω, για το θέμα του ελέγχου σε ό,τι αφορά τις γραμματείες. Οι γραμματείες είναι αυτές που μας υποστηρίζουν. Καλό λοιπόν είναι να υπάρχει μια άμεση όντως όχι μέσω των βουλευτών που έχουν πολλές αρμοδιότητες, πολλές δουλειές και το προλαβαίνουν. Νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε κατευθείαν τι θα πρέπει να γίνει. Αυτά νομίζω ότι είναι τα ερωτήματα και εγώ θα από πλευρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι. Oh, thought you would take so much more time. Α, νομίζω ότι θα απαντήσετε πολύ πιο αναλυτικά. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσω το λόγο σε ένα από τους ευρωβουλευτές, ακόμα μια φορά, στον κύριο Μαχτά. Για πολύ λίγο κύριε Μαχτά. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Οι καλεσμένοι μας δεν είναι εδώ για να συζητήσουμε ένα συγκεκριμένο θέμα. Ε, πάντως θέλω να σας πω ότι λυπάμαι που δεν απαντήσατε σε, στις ερωτήσεις μας. Δεν μιλάμε για απαγωγές παιδιών. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να σεβαστούμε δικαιώματα και των δύο γονιών. Γιατί από ό,τι φαίνεται η Γερμανία έχει το τεκμήλιο της ενοχής στη χώρα. Ε, ίσως θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε όταν περάσουμε στις αναφορές. Είπα προηγουμένω ότι αυτό για μας είναι θέμα και αρμοδιότητα των ομοσπονδιακών κρατηδίων. Δεν το, το ομοσπονδιακών κρατηδίων δεν είναι θέμα του ομοσπονδιακού κράτους, γι' αυτό ήταν και η απάντησή μου τόσο σύντομη. Δεν σας ικανοποιεί ενδεχομένω, αλλά υπάρχει αυτός ο σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων σε ό,τι αφορά το επίπεδο το ομοσπονδιακό και τα ομόσπονδα κρατήδια. Ευχαριστούμε. Να πω στους συναδέλφους και από τις δύο επιτροπές ότι η Επιτροπή της Bundestag μας έστειλε αναφορές και αναφορές ευρωπαϊκής διάστασης με χρήσιμα στοιχεία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα που είναι όντως αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μόνο το 2013 και το 2014 λάβαμε από την Bundestag 50 αναφορές, που δεν είναι λίγες, είναι πολλές. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν εθνικά κοινοβούλια που έχουν μια επιτροπή αναφορών και αυτή η συνεργασία θα μπορούσε να βελτιωθεί με κάποια κοινοβούλια. Προφανώς με την Bundestag είναι πάρα πολύ καλή και υπάρχουν και κοινοβούλια που δεν έχουν επίτροπε αναφορών, γιατί έχουν τελείω διαφορετική δομή. Παραδείγματο χάρη Σουηδία. Ίσως λοιπόν αυτή η θαυμάσια συνεργασία θα μπορούσε να μα εμπνεύσει. Θα μπορούσε να εμπνεύσει και άλλα εθνικά κοινοβούλια. Και τώρα με μεγάλη χαρά και έχοντα ακούσει τις δηλώσεις σας και τις προτάσεις για το μέλλον, για να βελτιώσουμε τη συνεργασία στα πλαίσια αυτού του δικτύου που υπάρχει στα πλαίσια του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή, μπορώ να περάσω στο επόμενο σημείο, κλείνοντας αυτό το σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το 5, για να αφορά 0954 κάθος 2011 από ένα γερμανό υπηκό MS για την άνηση μεταχείριση σε ό,τι αφορά την καταβολή διοδίων στο αυστριακό τούνελ Felbert Tower. Ο αναφέρον δεν είναι εδώ. Ίσως οι αναφέροντες παρακολουθούν στο σπίτι τους μέσω του ίντερνετ ή ο αναφέρον τέλο πάντων. Ε, κάθεται στο γκαναπέ του και παρακολουθεί άνετα-άνετα τις διαδικασίες. δεν θα δώσω το λόγο στον αναφέροντα, ε, ο οποίο δεν παρίσταται, αλλά στον κύριο Φρέντρικ Ράσμουσεν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Η αρχή τη μη διάκριση στο άρθρο 18 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια θεμελιώδη αρχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση οι διακρίσει σε βάση εθνικότητας είναι κάτι που απαγορεύεται με βάση την εφαρμογή των ε, συνθήκων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το καθεστώς των διοδίων ε, σε αυτή τη διασταύρωση παραβιάζει αυτή τη θεμελιώδη αρχή, γι' αυτό ε, δεν δίστασε να αναλάβει δράση εναντίον της Δημοκρατίας της Αυστρίας. Βάσει της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, άρθρο 18 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο λοιπόν αυτό απαγορεύει όχι μόνο την άμεση διάκριση βάσει εθνικότητας, υπηκότητας, αλλά και τις έμεσες διακρίσεις βάσει τόπου κατοικίας ή καταχώρησης ε, οχήματος, ταξινόμησης οχήματος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η Επιτροπή έστειλε ένα ε, ευρωπαϊκό πιλωτικό έγγραφο 2012 και επίσημη ανακοίνωση το 2013 ε, και γνωμοδότηση το 2014. Βάσει αυτής της διαδικασίας, μετά από τη διαδικασία, οι αυστραϊκές αρχές ε, υιοθέτησαν ένα νέο καθεστώς διοδίων για τα εμπορικά οχήματα και εμείς το σημειώνουμε. Έχει αντικατασταθεί το κριτήριο της ταξινόμησης ε, με ένα άλλο σύστημα εκπτώσεων για τα εισιτήρια πολλαπλής χρήση, που είναι διαθέσιμα για όλους όσοι θέλουν να διασχίσουν ε, ε, αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει λοιπόν διάκριση για τα εμπορικά οχήματα. Όμω οι αυστριακέ αρχέ δεν είναι κατευθυμένε να προσαρμόσουν το καθεστώ διοδίων σε ό,τι αφορά τα γιοταχή ή τα ελαφρά οχήματα. Έτσι η Επιτροπή θέλει, εξετάζει το ενδεχόμενο να παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πλήρης ε, εξαίρεση από το, ε, το καθεστώς διοδίων ε, στο Ανατολικό Τυρόλ είναι ένα δυσανάλογο μέτρο το οποίο δεν αιτιολογείται από άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντο. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε που ήσασταν τόσο σύντομο. Συγκεκριμένο και περιεκτικό. Λοιπόν, τώρα θα δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους. Σήμερα θα αναλάβω α, στη θέση του συναδέλφου Μπέκερ, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να παραβρεθεί σήμερα και θεωρώ ότι το θέμα των διοδίων είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και για τους Γερμανούς συναντέλφους και χαίρομαι που δραστηριοποιήθηκε το η Επιτροπή γιατί τίθεται και ένα θέμα με διακριτική μεταχείριση. Κατά τις δικές μου πληροφορίες, η Αυστρία στις 24 Νοεμβρίου 2014 Τροποποίησε το σύστημα του. Και έτσι έχω να, αποκτήσει, να μια ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι άλλαξε το σύστημα, αλλά όχι για τα φορτηγά. Άρα το θέμα που έθιξε ο αναφέρον, το θέμα της διακριτικής μεταχείρισης δηλαδή, σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά οχήματα, εξακολουθεί να παραμένει κρεμές από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. θα γίνει τώρα, θα αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι έχει δίκαιο αναφέρον, ότι πρόκειται για την κριτική μεταχείριση. όντω. κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, κάτι άλλαξε η Αυστρία, αλλά όχι για τα ιδιωτικά οχήματα. Τρίτον, τι θα πρέπει να γίνει λοιπόν εφ' εξής. Αυτή είναι η δική μου ερώτηση από πλευρά τη Επιτροπή. Η Πρόεδρο, θέλει κανεί άλλο να πάρει το λόγο για το θέμα αυτό. Όχι. τότε προτείνω να το χειριστούμε ως εξή. Εφόσον η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία παραβάση και όλο το θέμα έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Α, όχι, όχι ακόμα. Όχι, αλλά θα γίνει σύντομο αυτό. Οι αποφάσει. Ε, πρέπει να ληφθεί απόφαση, μάλλον, για να απευθυνθεί στο δικαστήριο υπόθεση. Εντάξει, αλλά έχει ξεκινήσει η δικασία παραβάση και η Επιτροπή το έχει αναλάβει τα αντισανάλογα μέτρα, αυτή η υπόθεση διακρίσεων. Η μοναδική απόφαση που μπορούμε εμείς να πάρουμε είναι να αποφασίσουμε να μην είναι ανοιχτή η αναφορά. Και έτσι και να ακολουθήσουμε, να περιμένουμε το ε, τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας παραβάση και την εκδίκαση υπόθεση στο δικαστήριο. Και βεβαίως ε, θα ενημερώσουμε και τον αναφέροντα. για να ξέρει και αυτός ποια θα είναι η διαδικασία από σήμερα. Εντάξει, ευχαριστώ. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη, τη 1281 κάθετος 2012 ε, του BR. Ε, διατάξεις ε, που απαγορεύουν τις εκτόσεις για φάρμακα που δίνονται σε ασθενείς στη Γερμανία. Και το ίδιο ισχύει και εδώ. Ο αναφέρον δεν είναι μαζί μας σήμερα. Ελπίζουμε να παρακολουθεί τη συζήτηση μέσω διαδικτύου. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στην Κάτια Φρέντριξ, εκ τη της Ευρωπαϊκής Ευχαριστώ. Η αναφορά αυτή αφορά την γερμανική νομοθεσία που πέρασε το 2012 Βάσει των νομικών διατάξεων προβλέπεται ότι η νομοθεσία τιμολόγησης στη Γερμανία αφορά και τα φάρμακα που εξαιρούνται ή μάλλον που παρέχονται από φαρμακεία έξω από τη Γερμανία σε Γερμανούς ασθενούς, ασθενείς. Ο αναφέρον ε, έχει παραπονωθεί ότι έλαβε ε, ε, φάρμακα από φαρμακείο εκτός Γερμανίας που δίνει όμως φάρμακα στη Γερμανία. Βάσει πληροφοριών που έχουμε λάβει, οι, επιτροπές, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ξεκίνησαν μια διαδικασία πιλωτική ε, ζητήσαμε πληροφορίες από τη Γερμανία, απάντησε η Γερμανία, ε, δεν θεωρούνται ικανοποιητικές οι απαντήσεις και έτσι στείλαμε επίσημη ε, ενημέρωση στη Γερμανία το 2013 και ζητήσαμε την αιτιολόγηση της νέας νομοθεσίας. Οι γερμανικές αρχές απάντησαν το 2014 με την τεκμηρίωση του μέτρου αυτού. Κατά τη γνώμη τους Υπάρχουν λόγοι που συνδέονται με την προστασία της δημόσιας υγείας ε, για την ε, επαρκή και σταθερή παροχή ιατροφαρμακευτικών προϊόντων σε όλη την επικράτεια. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή αξιολογεί τα επιχειρήματα της ε, Γερμανίας και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα αποφασιστεί εάν θα περάσουμε στο επόμενο βήμα. Ε, επίσης ακούσαμε ότι μπορεί να υπάρξει και παραπομπή από γερμανικό δικαστήριο που μπορεί να προωθήσει αυτά τα ζητήματα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να δούμε αν αφορούν ακριβώς τα ίδια ζητήματα. Μπορεί δηλαδή να μην το παραπέμψουμε εμείς ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά ένα εθνικό δικαστήριο. Οι συνάδελφοι τώρα έχουν το λόγο για να συμμετάσχουν.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 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για μια φοιτήτρια τελικά ε, γερμανικής ηθαγένειας που κάνει τις σπουδές της στην Ολλανδία και που την ίδια μεταχείριση για τα έξοδα μεταφοράς ε, στα δημόσια μέσα μεταφοράς όπως και οι Ολλανδοί ε, φοιτητές. Εμείς συμφωνούμε με την άποψη της ε, ε, φοιτήτρες αυτής. Είχαμε και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Η Κομισιόν βασίζει την αποφασή της ή μάλλον την άποψή της στο άρθρο 18 της ε, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Οδηγία 2004-38 άρθρο 24 που μιλά για τα δικαιώματα των ε, ατόμων που διαμένουν σε ένα άλλο κράτος μέλος. Η Κομισιόν ε, πήγε στο δικαστήριο πέρυσι, το Μάιο, και η υπόθεση έχει νούμερο ε, C233 14 ολοκλήρωσε τη διαδικασία, ολοκληρώθηκε η προκαταπτική διαδικασία. Θα πρέπει να δούμε πότε θα ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία, γιατί τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν με την άποψη της Κομισιόν, γιατί πιστεύει ότι αυτά είναι έξοδα ε, διαβίωσης. Ε, όμως, ε, κατά την άποψη της φοιτήτριας, ε, εδώ αυτά είναι έξοδα διαφορετικά, έχουν να κάνουν όχι με το κόστος ζωής, αλλά με τις σπουδέ τη. περιμένουμε λοιπόν να δούμε πότε θα γίνει η ακροματική διαδικασία, τι θα αποφασίσει το δικαστήριο και θα δούμε αν εμεί έχουμε δίκιο, τότε η φοιτήτρια αυτή, η αναφέρουσα, θα λύσει έτσι το πρόβλημά της, αν η Κομισιόν έχει δίκιο. Το λέω έχουν ε, οι συνάδελφοι, ο κύριο Γιάρ. Εμείς ε, για τους Γερμανούς συναδέλφους σήμερα Πρέπει να πούμε ότι τα πράγματα είναι λίγο απλά σήμερα σε ό,τι αφορά τι υποθέσει. Είναι σαφέ. Όσο είναι ανοιχτή η διαδικασία, τα είπε πάρα πολύ ωραία. Είναι, από πλευρά, είναι στην πλευρά του αναφέροντα, δεν συμφωνεί το κράτο μέλος. Προφανώς θα πρέπει να πάει στο δικαστήριο η υπόθεση και θα πρέπει να περιμένουμε. Θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά έως ότου έχουμε απάντηση. And I see nobody else. I guess... Δεν βλέπω κανέναν άλλον. Περιμένουμε λοιπόν ακόμα το, την απόφαση του δικαστηρίου. Ανοιχτή λοιπόν παραμένει η υπόθεση, η αναφορά. Κάτι άλλο δεν έχουμε να κάνουμε. Έχετε δίκιο, Πίτερ. Είναι και κάποιες ε, υποθέσεις που είναι απλές σήμερα. Και για να απευθυνθώ στους ε, εκπροσώπους ε, του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Μην πιστέψετε ότι το κάναμε επίτηδε για να κάνουμε εύκολη τη συνεδρίασή μα σήμερα και την επισκέψή σα. Συμβαίνει καμιά φορά. Και επίση, ε, κανονικά, πρέπει να σα πω ότι δεν έχουμε τόσε πολλέ παραπομπέ ε, στο ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τυχαίνει, τυχαίνει. Just a second. Λοιπόν, μόλι έλαβα το μήνυμα ότι ο επόμενος εκπρόσωπο τη Επιτροπή ε, είναι καθοδόν, γιατί και εμείς ε, έχουμε κινηθεί πολύ γρήγορα. Είμαστε πολύ μπροστά στο πρόγραμμά μα που δεν συμβαίνει συχνά. Συνήθω πολλοί συνάδελφοι θέλουν να παίρνουν το λόγο και δεν θέλουν να τον δώσουν πίσω. Επομένω, ε, συνήθω απλώ κοιτάζομαι απόγνωση το ρολόι. Σήμερα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, να σας κάνω εγώ μια εισαγωγή. Λοιπόν, 1071 του 2012, Bernard Kletzenbauer, ελπίζω να το λέω καλά, πείτε, Γερμανός ε, υπήκος για τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Είναι μία από τις αναφορές που μας έχουν παρμευθεί από εσάς στην Γερμανική Επιτροπή Αναφορών. Επομένω αυτό θα σας ενδιαφέρει ιδιαίτερως, υποθέτω. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι ο αναφέρον ζητά σε αυτήν την αναφορά την ε, κατάργηση ε, της ε, χρήση τέτοιων γενικά τροποποιημένων οργανισμών. Θεωρεί ότι θα χαθεί η βιοπικιλότητα εξαιτία αυτού και φοβάται ότι οι ε, γενικά τροποποιημένοι οργανισμοί και θα αλληλοδιασταυρωθούν με τα φυσικά, τα απλά φυτά και ότι τελικά θα καταναλώνουμε όλοι μόνο γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα επιλογής. Επίσης φοβάται ότι ε, ότι υπάρχει η δυνατότητα μονοπόλησης ε, των, των σπόρων και του φυτικού υλικού. Ε, η Επιτροπή ανέφερε ότι είχε λάβει την απόφαση να δώσει μεγαλύτερη ευχαίρεια στα κρατημέλη σε ό,τι αφορά τους αντιδοτημένου και εγκεκριμένου γενικά τροποποιημένου οργανισμού στην επικράτειά του. Αυτό είναι λοιπόν ε, το πλαίσιο τη υπόθεση. Να περιμένουμε τώρα την Επιτροπή για να μας εξηγήσει ακριβώς ε, τη δική της άποψη και αν έχουν επιπρόσθετες πληροφορίες από όσα σας ανέφερα εγώ. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να πάρει το λόγο, να μας πει κάτι, μια ιστορία, ένα ανέκδοτο. Λίγο να μας διασκεδάσει. Πολύ σπάνια συμβαίνει αυτό, επομένω ε, μην διστάσετε. Good, Mrs. Stanke. Please, the floor is yours. <laughs> Kommt jetzt keine Geschichte. Κυρία Στάνκε, όχι, θα σας πω ούτε ιστορία, το ανέκδοτο. Εγώ στην Επιτροπή μου ξέρω ποια είναι τα μέλη της Επιτροπής ε, και ξέρω ότι πίσω κάθονται οι επιμελείς υπάλληλοι. Εδώ δεν βλέπω ε, από τη σειρά 1-3 να υποθέσω ότι έχουμε τα μέλη της Επιτροπής, μετά έχουμε τους προσκεκλημένους και ακόμα πιο πίσω έχουμε τους πολίτες που ενδιαφέρονται. Έτσι έχει κατάσταση. Oh, that's a good question. The two... Καλή ερώτηση λέει ο Πρόεδρος. Οι δύο-τρεις πρώτες σειρές είναι για τα μέλη. Ύστερα, από αυτή την πλευρά εδώ στο δεξί έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά έχουμε και ένα μέλος που θέλει να κάτσει στην πλευρά του Συμβουλίου. Μετά έχουμε τον Bundestag, μετά τον Bundestag έχουμε τους αναφέροντες, οι οποίοι κανονικά έρχονται και κάθονται, εμπειρογνώμονες, βλέπω ε, εκπροσώπους ε, της υπηρεσίας χάραξη πολιτικής της νομικής υπηρεσίας, επίσης πάντα είναι εκπρόσωποι της νομικής υπηρεσίας εδώ πέρα. Έχουμε τα και άτομα από άλλε επιτροπέ. Και η στραπή, η πίσω ή η βοηθή των συναδέλφων. Από αυτή την πλευρά έχουμε όλα τα μέλη της γραμματείας. Και την Επιτροπή. Μία αίθουσα μεστή γνώσης και εμπειρίας. I am happy to, to be uh, the chairman of this committee. Χαίρομαι ιδιαίτερα που προεδρεύω την επιτροπή αυτή και πρέπει να σας πω, επειδή θέσατε το ερώτημα, ότι τα μέλη τη επιτροπή Αναφορών, μια και δεν είναι νομοθετική η εργασία τη Επιτροπή Αναφορών, αλλά μια επιτροπή που ασχολείται άμεσα με, τα, με τις ανησυχίες και τα προβλήματα των επιτρόπων, τα μέλη άλλων επιτροπών όπου υπάρχει νομοθετικό έργο, Είναι διαφορετική η φύση, ο χαρακτήρας της Επιτροπής μας αυτής. Okay. Okay, you know what? Let's let's cut the small talk now because now I'm happy. Ας σταματήσουμε όμως ε, τα διάφορα. Να σας ε, συστήσω την κυρία Ντροτή Αντρέ, η οποία είναι από την, Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας εξηγήσει και την Αναφορά 1071 του 2012. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας δώσετε την δυνατότητα να εκφραστούμε πάνω σε αυτή την ε, αναφορά, η οποία κατατέθηκε από τον κύριο Μπάουερ για τους ε, γάμα όμικρον. Έχουμε ήδη δώσει απαντήσεις θα σας κάνω μια περίληψη όλων των απαντήσεων που δώσαμε και, ενημέρωση, και μια ενημέρωση γιατί υπάρχουν εξελίξεις από την τελευταία υποβολή των γραπτών απαντήσεων της Κομισιόν. Καταρχάς, αυτό που θέλω να πω πρώτα απ' όλα είναι ότι έχουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο πλήρες που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο αυστηρά του κόσμου για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Αυτή η νομοθεσία λέει ότι για κάθε γαμματά όμικρον πριν τεθεί στην αγορά θα πρέπει να υποβάλλεται σε μία αξιολόγηση κινδύνου που γίνεται από την Αρχή Διατροφικής Ασφάλειας, την ΕΦΣΑ, που βρίσκεται στην Πάρμα και μία αξιολόγηση από τα κράτη-μέλη. Αυτή η αξιολόγηση γίνεται αναπερίπτωση για κάθε γαμματα και με βάση κάποια πρότυπα τα οποία είναι πολύ ψηλά ούτως ώστε να προστατεύσουμε την ανθρώπινη υγεία, τη ζωική υγεία και το περιβάλλον. Στην πράξη, για να αξιολόγησουμε τον κίνδυνο, ζητάμε από τον Ετούντα να μας δώσει μία σειρά από δεδομένα και αυτά τα δεδομένα ε, αναφέρονται σε κατευθυντήριες γραμμές που μας έδωσε η ΕΦΣΑ οι οποίες ε, γραμμές επικαιροποιήθηκαν σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική επίπτωση τελευταία φορά το 2010. Αυτές οι κατευθύνσεις γραμμές της ΕΦΣΑ απαιτούν ο ετών να δώσει στοιχεία για την ε, επιμονή, τη διεισδυτικότητα στα φυσικά διατήματα και οικοσυστήματα, τη πιθανή μεταφορά γονιδίων ε, των φυτών γαματάφω ομικρών προς συμβατά ή οποιαδήποτε άλλη περιβαλλοντική επίπτωση στους οργανισμούς στόχους και μη στόχους. Όλα αυτά είναι τα επιχειρήματα που περιγράφει ο Ετών και όλα αυτά τα στοιχεία τα εξετάζει η ΕΦΣΑ, σας διαβεβαιώ. Να προσθέσω ότι υιοθετήσαμε στις 13 Μαρτίου το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο υιοθέτησαν μια νέα νομοθεσία και σε αυτή τη νέα νομοθεσία που αφορά την καλλιέργεια των γάμων όμικρων υπάρχει μια δέσμευση από πλευρά κομισιών που προβλέπουν τα δύο θεσμικά όργανα, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, η Κομισιόν να επικαιροποιεί τις κατευθυντήρες γραμμές που είναι η βάση ούτω ώστε η ΕΦΣΑ και ο ΕΤΟΝ να υποβάλουν το φάκελο. Αυτό θα το κάνουμε το 2017 και η Κομισιόν ε, ασχολείται ήδη ο ετών ή οι ετούντες, όσοι υποβάλλουν τους φακέλους δηλαδή, έχουν την υποχρέωση επίσης να ασκούν και μια παρακολούθηση της ε, επίπτωσης των περιβάλλων των προϊόντων που σε αυτή τη στιγμή σε αυτά αγορά. Μιλάμε για τα σχέδια εποπτείας. Αυτά τα σχέδια εποπτείας υποβάλλονται στην Κομισιόν, στα κράτη-μέλη και στην ΕΦΣΑ που τα εξετάζει μπορεί να συμβεί η ΕΦΣΑ να ζητήσει από τον ετών να αλλάξει το σχέδιο παρακολούθησης ή εποπτείας και η Κομισιόν φυσικά δίνει μεγάλη προσοχή, μεγάλη σημασία σε αυτό. Συμφωνούμε με τον, με τον Ετούντα ότι πρέπει να υπάρχει μια ελευθερία για τον καταναλωτή να μπορεί να διαλέγει προϊόντα συμβατικά που προέρχονται από την βιολογική γεωργία ή προϊόντα γάματα φόμικρο. Και αυτή η επιλογή πρέπει να υπάρχει και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το επιβάλλουμε κάποια πράγματα του ετούντα. Αυτός ο στόχος υλοποιείται από την Κομισιόν στην οδηγία για τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν κανόνες συνύπαρξη, όπως λέγονται. Είναι μια δυνατότητα που έχουν τα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν βοηθάει στη διαδικασία αυτή υπό την έννοια ότι καθορίζει με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συνύπαρξης τις καλές πρακτικές που βοηθούν τα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα. Τα κράτη-μέλη αποτελούν, συμμετέχουν και σε αυτό το Γραφείο Συνύπαρξης των οργανισμών και δίνουμε μεγάλη σημασία στις εργασίες του γραφείου αυτού. Από την άλλη τώρα, η νέα οδηγία η οποία υιοθετήθηκε από τους δύο συνομοθέτες επιβάλλει ένα επιπλέον μέτρο για τη συνύπαρξη. Και ξέρω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, εάν σε ένα κράτος μέλος υπάρχει μια καλλιέργεια ενός γάμα ταφόμικρον και σε ένα άλλο κράτος μέλος δεν υπάρχει, το κράτος μέλος που καλλιεργεί τον γάμα ταφόμικρον είναι υποχρεωμένο να προβλέψει μέτρα διασυνοριακά απέναντι στο άλλο κράτος το οποίο δεν καλλιεργεί τον γενετικά τροποποιημένο οργανισμό. Είναι μια επιπλέον υποχρέωση που προσθέθηκε στην νομοθεσία για τους γάμα ταφόμικρον και θα τεθεί σε ισχύ το 2017 αυτό το στοιχείο. Είναι ένα επιπλέον στοιχείο που ενισχύει αυτές τις υποχρεώσεις συνύπαρξης για τα κράτη-μέλη που καλλιεργούν γενετικά τροποποιημένου οργανισμού. Η επιλογή, απ' την άλλη. Η επιλογή εξασφαλίζεται και από την ετικέτα, από την ε, επισήμαση. Υπάρχει υποχρεωτική αναφορά των ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Υπάρχει ένα κατόφλι απλώ, όπου πάνω από την οποία πρέπει να αναφέρεται η ύπαρξη των γάμματα φόμικρων. Ε, κάτω από αυτό δεν υπάρχει υποχρέωση να αναφέρεται στην ε, ετικέτα. Η υποχρέωση δηλαδή και η δυνατότητα επιλογής εξασφαλίζεται και μέσω της ετικετοθεσίας. Δεν απαγορεύεται τώρα τα κράτη-μέλη ή οι εμπορευόμενοι να δημιουργήσουν συστήματα ετικετοθεσίας χωρίς δάματα φόμικρον. Το βασικό είναι να μην αναγκάζουμε τον κατανοητή να κάνει λάθος. Σε αναφέρει, σε ό,τι αφορά σε ό,τι αφορά το θέμα των διπλωμάτων τεχνία, των αφαίρεων αφαίρων, δύσκολη λέξη να την προφέρουμε στα γαλλικά, Μπορεί. υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία για τα διπλώματα τεχνία, που εναρμονίζει τους εθνικούς νόμους ό,τι αφορά τα διπλώματα αυτά και οι ποικιλίε πόρων που αποτελούν αντικείμενο ένα άλλου είδους νομικού τρόπου προστασίας απαγορε... ε, εξαιρούνται από τη δυνατότητα προστασίας τους από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Σε ό,τι αφορά την ε, ανησυχία του αναφέροντα για το πιθανό μονοπόλιο ε, σπόρων από κάποιες μεγάλες εταιρείες. Πρέπει να σας πω ότι η νομοθεσία για τους σπόρους ε, δημιούργησε ένα σύστημα με σκοπό να εξασφαλίσουμε την ποικιλομορφία των ειδών, των ποικιλιών και μια δυνατότητα οι εταιρείε να φέρουν τα προϊόντα τους στην αγορά. Έχουμε δηλαδή διαφορετικού μεγέθους εταιρείε ε, στον κλάδο αυτό των σπόρων. Και υπάρχει μια μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2013, η οποία επιβεβαίωσε ότι στον τομέα των σπόρων υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις διότι αυτές οι επιχειρήσεις ήταν σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής αγοράς πόρων. Η διαδικασία έτσι, συγκέντρωσης α, της αγοράς στα χέρια κάποιων εταιριών φυσικά είναι σαφής, αλλά υπάρχουν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η παρουσία των μικρομέσων επιχειρήσεων μας καθησυχάζει. Κατα, ε, κατακλείδη, θα ήθελα να σας πω, η Κομισιόν πιστεύει ότι ο αναφέρον πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι ήσυχο ότι η Κομισιόν ασχολείται με την αποστολή που έχει, να εξασφαλίσει δηλαδή ότι οι εγκεκριμένοι γάμα όμικρον δεν δημιουργούν κίνδυνο για την υγεία και για το περιβάλλον, ούτε καν για τη βιοπικιλότητα. Και να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει επιλογή για τον Ευρωπαίο καταναλωτή μέσω της επισήμασης, της αναφοράς δηλαδή των οργανισμών που είναι γενετικά τροποποιημένοι. Αυτά ήθελα να πω κυρία Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ. Τώρα το, το λέω έχουν οι συνάδελφοι. Η κυρία Σακοράφα. Και συνεχεία η κυρία Εύη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε να επισημάνω κάτι γενικά για την Επιτροπή και τον τρόπο δουλειάς της και τα αποτελέσματά της. Όπως έχω ξαναπεί την προηγούμενη φορά στην Επιτροπή, είναι αυτή η Επιτροπή το τελευταίο καταφύγιο των Ευρωπαίων, ε, αν θέλετε, πολιτών όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Από τη στιγμή λοιπόν που κάνουμε παραδεκτή μια αναφορά, σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε το βάσιμο των ανησυχιών των ανθρώπων αυτών και των καταγγελιών, των παραπώνων τους, γενικά δηλαδή του περιεχομένου των αναφορών που κάνουν. Και ο στόχος μας είναι με την παρέμβαση και τις ενέργειές μας να θεραπεύσουμε τις ε, επιτρέψτε μου να επαναλάβω αποδεκτές παραλήψεις και στρεβλώσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας μέχρι τώρα προκαλώντας βεβαίως μέσα από αυτή τη διαδικασία τις σχετικές νομοθεσίες και τις απαραίτητες οδηγίες ή αν θέλετε και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Αν και στην ε, αναφορά που συζητάμε φαίνεται ότι με τις ε, οδηγίες που έχουν εκδοθεί καλύπτονται και απαντούνται όλες οι ανησυχίες του αναφέροντος, θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω ότι η ανάθεση της ευθύνης σε κάθε κράτος ξεχωριστά, κατά πρώτον, είναι υπεκφυγή από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις ευθύνες της και δεύτερον, με δεδομένο ότι η φύση δεν ορίζει γεωγραφικά σύνορα, ουσιαστικά απαντάμε στις ανησυχίες του αναφέροντας, τις οποίες κάνουμε βεβαίως παραδεκτές, όπως φαίνεται και από το σχετικό έγγραφο, ε, δηλαδή ασπαζόμαστε τις ανησυχίες του, νομοθετώντας για την κυκλοφορία των εντόμων, του νερού, του αέρα κτλ. Ουσιαστικά δηλαδή οι ανησυχίες των πολιτών και του αναφέροντος συνεχίζουν να είναι πραγματικές και μετά τις οδηγίες. Δεν είμαι έτοιμη αυτή τη στιγμή να προτείνω σε ποιε παραπέρα ενέργειε θα μπορούσε να προβεί η Επιτροπή ώστε να υποχρεώσει σε μια ουσιαστική συμμόρφωση τη νομοθεσία, αλλά εκτιμώ ότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα, παρόλο που τυπικά η αναφορά δεν έχει λόγο να μείνει ανοιχτή, θα πρότεινα να μείνει ανοιχτή ώστε να αποτελέσει βάση προβληματισμού στην κατεύθυνση που ανέφερα παραπάνω. Επειδή λοιπόν εκτιμώ το γεγονός ότι η Επιτροπή και διάθεση δείχνει και αποφασιστικότητα να μπαίνει στην ουσία των ζητημάτων, πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι το συγκεκριμένο, να επεξεργαστούμε μια παραπέρα παρέμβαση ώστε να καταλήξουμε στην ουσιαστική αντιμετώπιση των ανησυχιών όλων των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. And Κυρία Εύη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Παρά τις διαβεβαιώσεις που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ θέλω να υποστηρίξω τις ανησυχίες που εκφράζει ο αναφέρον. Γιατί παρά τη νέα αναθεώρηση της ε, παλιάς οδηγίας 18 ε, του 2001 που δίνουν τη ε, δυνατότητα στα κράτη-μέλη να απαγορεύσουν την καλλιέργεια στην επικράτειά τους. Υπάρχει μια σειρά από δράσεις, το λεγόμενο opting out, δηλαδή τη δυνατότητα να εξαιρέσουμε την επικράτειά μας από την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Παρ' όλα αυτά, αυτό το μοντέλο, αυτές οι δράσεις επαναλαμβάνονται και για τις τροφές ε, με βάση τους γάμα τα Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για την καλλιέργεια πια, αλλά και για τα τρόφιμα. Είναι ένα προηγούμενο που, που αποδυναμώνει το κράτος μέλος, νομίζω. Γιατί τη στιγμή που το κράτος μέλος απαγορεύει την καλλιέργεια ή την το εμπόριο για την κατανάλωση στο εσωτερικό των συνόρων του, των γαματαφόμικρων, βρίσκεται σε αδύναμη νομική θέση. Γιατί μπορεί να υπάρξει μια προσφυγή μιας μεγάλης εταιρείας στο πάνελ του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Και το κράτος αυτό πραγματικά είναι ευάλωτο. Και αν προσφύγει εναντίον του μια μεγάλη εταιρεία, τότε το πράγμα συγκεκριμενοποιείται αντιμετωπίζει μια απειλή. Το να δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη το να απαγορεύουν εντελώς την χρήση των γάμα όμικρων, νομίζω είναι ένας τρόπος ε, για να πετάξει το μπαλάκι από το γήπεδό της Κομισιόν, να το ξεφορτωθεί από τους ώμους της και την πλάτη της και να αφήσει τα κράτη-μέλη μόνα τους να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε, μια ενδεχόμενη προσφυγή που θα γίνει ενώπιον του πάνελ του α, Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η ΕΦΣΑ που είναι ο οργανισμός ο οποίος αποφαίνεται για την ασφάλεια των ε, προϊόντων διατροφής και εγκρίνει τη θέση στο εμπόριο και την καλλιέργεια των γάμα ομικρών, μην ξεχνάμε ότι είχε την ε, είχε διάφορες σχέσεις μεταξύ ε, επιστημόνων, με εταιρείε και τα με τις με τις ε, πολυεθνικές της ε, βιοτεχνολογίας που του δίνουν. Δηλαδή οι εταιρείε αυτές ε, δίνουν στοιχεία στην ΕΦΣΑ με βάση τα οποία η ΕΦΣΑ δίνει τις εγκρίσεις αυτές, τις άδειε στα προϊόντα. Προσοχή, προσοχή λοιπόν. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά για να μην ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι το να συζητάμε αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κύριος Βασισόφσκι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι η τρίτη μου κοινοβουλευτική εκθετία και επικεντρώνομαι κυρίως στις δραστηριότητες μου στην Επιτροπή Γεωργίας. Επομένω τα γνωρίζω όλα αυτά, αυτή τη συζήτηση για τους γάμματα φόμικρων. Πριν από 10 χρόνια, όταν όλος ο κόσμος έλεγε ότι οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί είναι ε, απειλή, υπήρχαν κάποιοι τρελοί εντό αγωγικών που πήγαιναν ενάντια στην επιστήμη. Όμως μεταξύ, μάθαμε πολλά για την απειλή, ε, τον κίνδυνο που ενέχει η καλλιέργεια και χρήση των γάματα όμικρων, για την υγεία, την ασφάλεια, αλλά και για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδο, αναφέρθηκε και εδώ και υπάρχει συμβιβασμός σε εθνικό επίπεδο ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει αν θα δεχθεί ε, τις καλλιέργειες γάμματα φόμικρον ή όχι. Βέβαια αυτό δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Γιατί ορισμένες φορές είναι δύσκολο να, το, να ελέγξει κανείς την κατάσταση, υπάρχει παράνομη καλλιέργεια γάμματα φόμικρον. Εγώ προσωπικά χαίρομαι που έχει καταβληθεί αυτή η αναφορά. Ξέρω και χαίρομαι μάλλον που υπάρχει ακόμα ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα συζητήσουμε στην Ευρώπη γιατί είναι και θέμα επιλογής τύπου γεωργίας. Αν αφήναμε την, επιτρέπαμε την καλλιέργεια γάμματα αφόμικρων ε, στην Ευρώπη και αν το κάνουμε αυτό στο μέλλον θα καταλήξουμε να έχουμε το μεγαλυντικό πρότυπο γεωργίας και στην Ευρώπη. Γιατί οι ε, γάμματα αφόμικρων πρέπει να καλλιεργούνται σε τεράστιες εκτάσεις και έτσι θα τεθεί ένα τέλος στην οικογενειακή γεωργία, τους μικρούς δηλαδή γεωργούς. Εγώ είμαι κατά των γάματα ταφόμικρων, πρέπει να έχουμε πλήρη απαγόρευση τους ε, στην Ευρώπη. Έχουμε εύρωστα επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν ότι ε, αποτελούν κίνδυνο γαματοφόμικρον στην ε, παραδοσιακή βιολογική καλλιέργεια αλλά και στην ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ζώων. Ευχαριστώ. Κύριος Πιτεριάς also aus meiner Sicht... Äh, από δική μου πλευρά ε, είναι πολύ καλή αυτή η αναφορά από το 2012 και μπορούμε λοιπόν την αναφορά αυτή να τη θεωρήσουμε και πάρα πολύ επιτυχημένη γιατί πολλά πολιτικά κίνητρα έδωσε και έθεσε. Από το 2012 μέχρι σήμερα Πολλές νομοθετικές αλλαγέ έγιναν, αυτό το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο συνάδελφο από την Επιτροπή Γεωργίας. Πολύ σωστά τα παρουσίασαν όλα αυτά. Τα προβλήματα τα οποία ακούσαμε, αξιολόγηση κινδύνου έγινε και επίση ε, συμφωνήσαμε αν καταλήξει στο συμπέρασμα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλιση Υπήρξε μια ιδιαίτερη κατάσταση πριν από κάποιο καιρό γιατί δημιουργήθηκε αυτή η Ευρωπαϊκή Συμβασμός, ε, ο κανονισμό αυτός. Αυτό πιστεύω ότι αποτυπώνει και αντικατροπτρίζει την αλήθεια σε ό,τι αφορά το συμβασμό, ο οποίος πλέον υπάρχει. Μία λοιπόν ε, προϋπόθεση πληρείται το θέμα της ευρεσιτεχνίας τώρα. Χαίρομαι που σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη δεν ε, επιτρέπουν ε, κατοχύρωση μέσω ευρωστεχνίας ε, τέτοιων ζώντων οργανισμών για ζώντους οργανισμούς φυτά ότι αποφάνθηκε έτσι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε μία απόπειρα τέτοια αναφέροντας ότι θέλουμε να κατοχυρώσουμε με βρεστεχνία την τεχνική διαδικασία και έτσι μέσω της τεχνικής διαδικασίας ε, κατοχυρώνονταν και το αποτέλεσμα, το φυτό. Αυτή η απόπειρα μπορέσαμε να αντισταθούμε σε αυτήν. Και αυτό λοιπόν εκπληρώνεται και πληρείται ω όρο. Φυσικά πρόκειται για τονισμό. Εγώ και οι πιο πολλοί εδώ στην Επιτροπή, τα κρατημέλη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θέλουμε να υπάρχουν ευρεσιτεχνία σε ε, ζώα, φυτά, ζώντου οργανισμού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό λοιπόν πληρείται ω όρο. Επίλογη ελευθερία επιλογής για τους καλλιεργητές. Εδώ να προσέξουμε. Δεν πρέπει να μπλέξουμε τους ε, σπόρους, την τεχνολογία των σπόρων και τις γενετικούς οργανισμούς, τροποποιημένους οργανισμούς. Το πιο σημαντικό όπλο του καλλιεργητή, του αγρότη, είναι η επιλογή, η ελευθερία επιλογής. Το φυτό το οποίο έχει επιλέξει να καλλιεργήσει μπορεί να αναπαραχθεί μόνο του. Κάθε λοιπόν καλλιεργητής θα πρέπει να έχει δικαίωμα για το επόμενο έτος. Και η νομοθεσία για τους πόρους ε, η ευρωπαϊκή είναι πάντα στην πλευρά του αγρότη, του καλλιεργητή. Αυτό θα πρέπει να μείνει έτσι. Στο παγκόσμιο επίπεδο, σε διεθνέ επίπεδο, υπάρχουν κακά παραδείγματα. Γιατί αν ε, ω καλλιεργητή υποχρεώνουμε κάθε χρόνο να αγοράζω καινούριου πόρου, εξαρτάμε από, τον, ε, από την αγορά. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Θα πρέπει να υπάρξει η ελευθερία επιλογή του σπόρου τη ε, καλλιεργία. Δεν θα πρέπει να υπάρξει μονοπόλιο από αυτήν την άποψη αυτή. Να ανοίξω εδώ μια παρένθεση και να πω το εξή. Να προσέξουμε σε ό,τι αφορά του ε, σπόρου και την παραγωγή σπόρων. Να τα βγάλει πέρα η μικρομεσαία τάξη να μην μείνουν ε, μόνο λίγοι μεγάλοι σε όλο τον κόσμο σε ό,τι αφορά την παραγωγή σπόρων. Άρα, συνολικά, εγώ θα μπορούσα να πω ότι και να φανταστώ ότι θα κλείσουμε την αναφορά. Έχει κινηθεί πολύ η κατάσταση, πληρούνται οι όροι και προποθέσει. Φυσικά, ε, εξελίσσεται η κατάσταση, η ζωή προχωράει, θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσει. σε ό,τι αφορά τα θέματα της ευρεσιτεχνίας στους ζώντους οργανισμούς, σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, ελευθερίας επιλογής του καλλιεργητή, νομίζω ότι τα πράγματα πήγαιναν σε καλή κατάσταση από το 2012 και μετά. Να ακούσω τι έχουν να, πει, να πούν και οι άλλοι συνάδελφοι, κατά πόσο έχουν αμφιβολίες, αλλά εγώ είμαι μάλλον ικανοποιημένος. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο για αυτό το θέμα. Εντάξει, τότε πρέπει εγώ να κάνω τη σύνοψη. Είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι ήταν ε, ιδιαίτερα εμπιστευμένη η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε μεγάλη λεπτομέρεια μας ε, ανέλησε η Επιτροπή τι ακριβώς έχει γίνει από την υποβολή της ε, αναφοράς 2012. Και ο Πίτερ αυτό ανέφερε, ανέφερε κάποια στοιχεία δεν νομίζω ότι αυτή η συγκεκριμένη αναφορά θα πρέπει να αποτελέσει σύμβολο της μάχης κατά των γαματαφόμικρων γενικά. Είναι τόσο ευρύ αυτό το ζήτημα που πρέπει όλοι από κοινού να παρακολουθούμε τι συμβαίνει σε αυτό το πεδίο. Όμως νομίζω ότι τα σημεία προβληματισμού αυτού του κυρίου, του αναφέροντος, έχουν αντιμετωπιστεί και απαντηθεί καταλήλω. Νομίζω λοιπόν ότι για τη συγκεκριμένη αναφορά μπορούμε να την κλείσουμε και να παρακολουθήσουμε γενικά το ζήτημα και τη συζήτηση. Όμω θα πρέπει να δώσουμε γραπτό, στον αναφέροντα και αυτή την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είτε εκ μέρου σας, είτε μπορείτε να το κάνετε εσείς, αλλά θα θέλαμε και εμείς ένα γραπτό αντίγραφο της απάντησής σας. Αυτό νομίζω ότι είναι μια καλή συμβαστική λύση. Δηλαδή να προωθήσουμε όλες τις ε, λεπτομέρειες της ενημέρωσης αυτής προς τον αναφέροντα και να τον ε, ενημερώσουμε και να τον διαβεβαιώσουμε μάλλον ότι αυτή η συζήτηση δεν έχει τέλος και συνεχίζεται πάντα. Αυτά ήθελα εγώ να προτείνω. Δεν ξέρω αν έχουν και συνάδελφοι κάτι να πούν. Could we do that? Συμφωνείτε? Διαφωνεί κάποιος? Ωραία. That's good. Thank you. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λοιπόν ευρεία συνένεση για αυτό το θέμα και χαίρομαι και πάλι με τα χαρά να στραφώ στους συναδέλφους από την Bundestag να σας πω ότι τους ζυγούς λύσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα και προσβλέπουμε να ανταλλάξουμε απόψεις σε, σε κάποια άλλη περίσταση. Για τους υπόλοιπους, τουλάχιστον τους συντονιστές, τα λέμε στις 5 παρατέταρτο ακριβώς.